Pan Przewodniczący! Good afternoon. I'm sorry for being a bit... Καλησπέρα σας και ευχαριστώ συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω. Είχαμε όμως ένα διαδικαστικό ζήτημα. Όπως θα θυμάστε ίσως, είχε υποβληθεί έτοιμα από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε σχέση με τη συζήτηση για τον Γκουαντάναμο Είχαμε φτάσει στο δεύτερο σημείο του θέματος αυτού. Συνεχίστε λοιπόν στις συνεδρίασεις. Έχει υποβληθεί από τον κύριο Μποργκέτσιο έτοιμα για μια προσωπική δήλωση. Σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Ξεκινούμε με την προσωπική δήλωση του κύριου Μποργέτσιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα διαβάσω την επιστολή που απέστειλα σήμερα το πρωί στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τις δηλώσεις που εκφράσατε στην έναρξη της Συνόδου την Δευτέρα 20 ε, Μαΐου 2013, πρέπει να πω ότι ε, εκφραστήκατε για την Υπουργό με τρόπο αρκετά σαρκαστικό, ε, για την Υπουργό Κέζεφ και θέλω να τη ζητήσω προσωπικά συγγνώμη εγώ δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν με τα λόγια μου και ευχαρίστω να τα αποσαφηνίσω, γιατί οι πραγματικέ μου προθέσει μπορεί να έγιναν αντιληπτέ ω ε, απόπειρα προσβολή κατά μια προσωπικότητα που αξίζει το σεβασμό μας και είναι και γυναίκα βεβαίω. Λυπούμε ιδιαίτερα εάν οι εκφράσεις μου φάνηκαν ε, επιθετικές και περισσότερο είχαν να κάνουν με την πολιτική μετανάστευση και την αιτιολόγηση της δικής μου τοποθέτησης. Ουσιαστικά, ο υπουργό δεν συμφωνούσε και είχε εκφράσει διαφορετικές απόψεις από τη ομάδα μας, η Ευρώπη της Δημοκρατίας και Ελευθερίας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μποργκέτσιο. Και επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι έχω λάβει αίτημα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο δυνάμει του άρθρου 177 παράγραφος 1 του κανονισμού για αναβολή τη συζητήσεω για το Γουαντάναμο που προβλεπόταν για την πέμπτη το απόγευμα. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν θέλει τον λόγο ο κύριο τώρα. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί ε, κατέθεσα αυτό το αίτημα εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας για να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε τη συμφωνία της Ολομέλειας